Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Nous reprenons nos travaux. J'indique que notre... Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε εργασίες μας. Έχει κατά τροποποιηθεί και σήμερα το πρωί για λόγους χρονοδιαγράμματο δεν μπορούμε να ακούσουμε την Κλέρ αναφορικά με τον έλεγχο του προπολογισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ από τον προπολογισμό της Ένωσης και δέχτηκε να μας παρουσιάσει την έκθεσή της το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Δίνω το λόγο τώρα στον κ. Γκάγερ για να μας μιλήσει σχετικά με τους κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το έργο αυτό που μου είχε ανατεθεί. Επρόκειτο για τροποποίηση βασικού κανονισμού του οργανισμού ΕΑΣΑ. Το θέμα μου άλλωστε είναι κοινή κανόνη των στον τομέα τη πολιτική αεροπορία και σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια τη Αεροπορία. Αυτό ο κανονισμό είναι μέρο τη στρατηγική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που θεσπίστηκε από το 2015, δηλαδή η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της ΕΑΣΑ που συναποτελεί μέρος του συνολικού πακέτου. Η διάρθρωση του προϋπολογισμού της ΕΑΣΑ έχει περίπου ως εξής. Ένα μέγα μέρος χρηματοδοτείται από εισφορές και τέλη της ε, Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Βιομηχανίας για πιστοποιήσεις και άλλα σχετικά, βιομηχανίες κατασκευής αεροσκαφών δηλαδή, άλλο μέρος από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ένα πολύ μικρό μέρος από τις φορές τρίτων χωρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι στον προϋπολογισμό της ΆΣΑ υπάρχει μια διπλή δομή και σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση του προϋπολογισμού αλλά και σε ό,τι αφορά το οργανόγραμμά της. Εκεί μπορούν να γίνουν και εξοικονομήσεις βεβαίως εάν δηλαδή μπορέσει να ισχύσει μια κοινή προσέγγιση για τον προϋπολογισμό, κάτι το οποίο προτείνω άλλωστε. Αυτό θα διευκολύνει την ε, διοίκηση, διαχείριση. Θα συμβάλλει επίσης, διότι κατά την γνώμη μου χρειάζεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα καθήκοντα του οργανισμού αυτού που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία και σε εκείνα που χρηματοδοτούνται από δημόσιο προπολογισμό ή που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται. Αλλά διαχωρισμός ο οποίο δεν μπορεί να είναι απόλυτος. Εξηγήστε μου, για παράδειγμα, πώς θα χρηματοδοτείται ο μισθός του διευθυντού της ΕΑΣΑ. Όπως είπα, εν μέρη χρηματοδοτείται η ΕΑΣΑ από εισφορές και τέλη, πιστοποιήσεις κλπ της βιομηχανίας, άλλο μέρος από τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Ειδικότερα λοιπόν για προσωπικό και διοικητικά μέσα στον ίδιο τον οργανισμό θα είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς ότι αυτό το τμήμα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα τέλη, αυτό πρέπει να την χάνει δημόσια χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Επομένως, το ύψος των τελών υπολογίζεται σε βάση κάποιων αξιόπιστων στοιχείων, αλλά δεν μπορεί να είναι υπολογισμένο μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ. Ούτε νομίζω άλλωστε ότι είναι και το κρίσιμο στοιχείο, διότι μίλησα με προσώπους της ε, Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Βιομηχανίας και το μήνυμα που μετέφεραν ήταν ότι κρίσιμο για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία αεροναυπηγική βιομηχανία δεν είναι το ύψος των τελών. Κρίσιμο είναι η ταχύτητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, διότι από αυτή την ταχύτητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προκύπτει, απορρέει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής αεροπορικής βιομηχανίας. Αν λοιπόν μπορέσουμε να επιλέξουμε την προσέγγιση που ανέφερα πριν, θα γίνει άσα ένας οργανισμός που θα επιτρέπει την τοποθέτηση του προσωπικού εκεί όπου πραγματικά είναι αναγκαίο και όχι αναλόγως με το από πού χρηματοδοτείται, δηλαδή αν η χρηματοδότηση είναι δημόσια, ιδιωτική και ούτω καθεξής. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει άρα είναι η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα με την οποία ο οργανισμός ΕΑΣΑ μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και η ενδεχόμενη δυνατότητα αύξηση της ταχύτητας αυτής. Και με την επιλογή που προτείνω νομίζω θα τα καταφέρουμε. Σήμερα έχουμε διαχωρισμό, έχουμε διαίρεση του προσωπικού ανάμεσα σε αυτούς που εργάζονται για τη βιομηχανία και αμείβονται από τέλη αυτής, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει μείωση 5% στο προσωπικό, δεν, δεν αποτρέπει δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει μείωση κατά 5% του προσωπικού του ΕΑΣΑ. Κάτι το οποίο βρίσκω άδικο, διότι το προσωπικό το οποίο χρηματοδοτείται από τις υπηρεσίες που παρέχονται στην βιομηχανία δεν θα πρέπει να υποστεί τέτοια περικοπή, διότι οι υπηρεσίες που παρέχονται ωφελούν την βιομηχανία. Έτσι και αν επιλογεί, και αν δηλαδή ο ενιαίος προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να περικοπεί το προσωπικό αυτό διότι στόχος της ΕΑΣΑ και του μέρους αυτού του προσωπικού της είναι να παρέχει υπηρεσία στη βιομηχανία. Κάτι που με απασχολεί ακόμη και που είναι κάπως δυσάρεστο, σας το λέω ειλικρινά, ως πολίτη της Ομοσπονδιακής Γερμανίας είναι το γεγονός ότι η ΕΑΣΑ δεν έχει ακόμα συμφωνήσει οριστικά για την έδρα της με την ε, γερμανική κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα για τον οργανισμό Frontex και το πολωνικό κράτος. Ο ΕΑΣΑ που είναι και παλαιότερος οργανισμός από τον Frontex τελικά εξακολουθεί να πάσχει από αυτό το δεινό. Και γι' αυτό περιλαμβάνω στη γνωμοδότησή μου το ότι αναμένουμε η συμφωνία μεταξύ ΕΑΣΑ και Ομοσπονδιακής Γερμανίας να λάβει επιτέλους τελική μορφή σχετικά με την έδρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ τον κύριο Γκάια και βεβαίως στηρίζουμε την Γερμανία να υπογράψει τη σύμβαση για την έδρα με την ΕΑΣΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω σαν σκιώδη εισηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ. Θέλω να υπογραμμίσω κάποια σημεία. Καταρχήν, πρέπει όταν καθορίζουμε τον προϋπολογισμό να μην ξεχνάμε ότι οι διαφορετικές υπηρεσίες έχουν διαφορετικό ρόλο και καθήκοντα. Και βάσει αυτού γίνεται και η ανάλυση. Κοιτώ λοιπόν τις τροπολογίες και εάν πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση 100% από τον ιδιωτικό τομέα, έχω κάποιες ερωτήσεις. Πώς είναι δυνατόν τα τέλη, τα ιδιωτικά, η ιδιωτική χρηματοδότηση να καλύψει κάποιες ε, αρμοδιότητες ε, που είναι καθαρά του δημόσιου τομέα, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν αυτό να καλυφθεί μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, από ιδιωτική χρηματοδότηση. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο προκύπτει. Διότι θα υπάρξει χάος εάν προσπαθήσουμε να περάσουμε από το σημερινό διαρθρωμένο σύστημα σε ένα ε, σύστημα 100% ιδιωτικής χρηματοδότησης. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο το ακούμε από πολλές πλευρές, όχι μόνο από πλευράς ε, ελέγχου του προπολογισμού. Είναι το θέμα των ε, αντικρώμενων συμφερόντων. Και εγώ θέλω να το θέσω αυτό το θέμα. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή ε, προτείνει να λάβουμε υπόψη μας και τα συμφέροντα αυτά. Εάν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε την πρόταση της Επιτροπής, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε άλλου είδους ε, δυσκολίες και βάρη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ένα τελευταίο σημείο. Αν ζητήσουμε την ίδια την υπηρεσία, θα σας απαντήσουν ότι κάτι τέτοιο σίγουρα δεν θα βοηθήσει ούτε και για τα λογιστικά. Κύριε Γκάιρ, δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί εδώ προτείνουμε να αλλάξουμε το σύστημα που υπάρχει και λειτουργεί και να κατευθυνθούμε προς κάτι τελείως διαφορετικό. Ποιος ζητάει το λόγο? Η κυρία Χολμάιερ. Κύριε Πρόεδρε, εσείς και εσείς κύριε Γκάιερ, εσύ που παρακολουθείς τόσο προσεκτικά τα δρόμενα της ΕΑΣΑ. Ανησυχώ κάπως ότι προσπαθώντας να εφαρμόσουμε ένα γενικό μοντέλο σε όλους αυτούς τους οργανισμούς μπορεί να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Οργανισμοί όπως Eurojust, Europol, εκεί δεν μπορεί τίποτε να είναι fee paid, να πληρώνεται δηλαδή από τέλη ή εισφορές. Όλα πληρώνονται από τον κοινοτικό προπολογισμό. Στην ΕΑΣΑ τα πράγματα είναι ξεχωρισμένα. Όταν πρόκειται για πιστοποίηση, έχει απόλυτο δίκιο ότι εκεί είναι ζήτημα ταχύτητας. Όμως, εξαρτάται και από το ύψος των τελών. Και εδώ δεν μιλούμε μόνο για τις μεγάλες βιομηχανίες, διότι έχουμε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ύψος των τελών αυτών, Όπω μπορεί εντελώ αυτονόητα η μεγάλη βιομηχανία. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν λοιπόν πολύ σημαντικότερε δυσκολίες. Στον τομέα δε αυτών υπάρχει πλήθος, ξαναλέω, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είναι μονάχα η Airbus και η Boeing που έρχονται να ζητήσουν πιστοποιήσει για τα προϊόντα τους, υπάρχουν και πολλές, πάρα πολλέ μικρές ή και μεσαίες επιχειρήσει. Βρίσκω ιδιαίτερα προβληματικό να προχωρήσουμε σε μια χρηματοδότηση που να είναι εξασφαλισμένη μόνο στη βάση τελών που θα καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις. Δεύτερο, νομίζω ότι υπάρχει ένα μέρος του ΕΑΣΑ που πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε βιομηχανική επιρροή. Βεβαίως θα συνομιλεί με τη βιομηχανία και συνομιλούμε και εμείς, αλλά για θέματα ασφαλείας πρέπει ασφαλώς να είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι από την βιομηχανία. Ασφαλώς και η βιομηχανία θα πει τη γνώμη της. Αλλά πρέπει η ανεξαρτησία του θεσμού να είναι απόλυτα εξασφαλισμένη. Για θέματα ασφαλείας, επαναλαμβάνω, δεν επιτρέπεται αυτά να χρηματοδοτούνται από εισφορές, τέλη κλπ. Όπως κάνουμε και για τις αστυνομικές δυνάμεις. Διότι μάλιστα αυτό μπορεί να οδηγήσει και στην αποφυγή λήψης μέτρων που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικά, χρήσιμα και αναγκαία δεν προκύπτουν αυτομάτως συγκρούσεις συμφερόντων. Νομίζω ότι υπάρχουν τομείς δραστηριότητας της ΕΑΣΑ ή του ΕΑΣΑ που πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερα από οποιαδήποτε χρηματοδότηση στη βάση τελών. Πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τρίτο, πάντα στο ίδιο πλαίσιο, τα τέλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν τομεί του γενικού προϋπολογισμού. Τα τέλη έχουν πάντοτε ειδικό χαρακτήρα, δηλαδή καταβάλλονται για να καλύψουν το κόστος, για παράδειγμα, μιας πιστοποίησης. Και άποψη, από άποψη συνταγματική, τουλάχιστον από την άποψη της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Βρετανικής νομολογίας, αυτά απαγορεύουν να μετατραπούν τα τέλη σε κρυμμένη φορολόγηση και να χρησιμοποιηθούν επομένω για σκοπού αλότριου από αυτού για του οποίου προβλέπονται από τον νόμο. Ήδη δηλαδή το δίκαιο δεν το επιτρέπει αυτό. Άρα χρειάζεται να ε, προχωρήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά, να συζητήσουμε πολύ προσεκτικά το τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να αποφύγουμε να μπούμε σε ύδατα τα οποία ενδεχομένως νομικά είναι εντελώ αβέβαια. Και επαναλαμβάνω, είδαμε και τελευταία το τραγικό ατύχημα της Αιγυπτέα Εάν πραγματικά αποδειχτεί ότι στην τουαλέτα του αεροσκάφους είχε τοποθετηθεί βόμβα, κάτι για το οποίο φαίνεται να συνηγορεί η κατάσταση των ανθρώπινων μελών που βρίσκονται στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των αεροσκαφών, ποιε είναι οι προποθέσει, θα αντιμετωπίσουμε ασφαλώ καινούρια προβλήματα, διότι είναι η δεύτερη βόμβα που τοποθετήθηκε σε αεροσκάφο και η οποία εξεράγει προφανώς, προφανώς από εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων που ε, προσφέρουν τα αναλώσιμα στα αεροσκάφη και ούτω καθεξής. Αυτά τα πράγματα πρέπει να καταβάλλονται, δηλαδή οι έρευνες και οι διατάξεις ασφάλειας των αεροσκαφών πρέπει να πληρώνονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για να καταλήξουμε και στο του δυνατό αποτέλεσμα. Πάντως ευχαριστώ για την θετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφός μας τώρα, ο Μπενίτου Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ουσιώδης ηγητής ε, από την ΚΟΕ, να εκφράσω την άποψή μου επί της εκθέσεως. Είναι προφανές ότι ο τομέας ε, της ε, πολιτικής αεροπορίας είναι ένας τομέας το οποίο προβλέπεται μια περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις προκλήσεις που έχουν προκύψει με έναν τρόπο αποτελεσματικό, αλλά θα πρέπει να, ε, δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της ε, ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ε, πιστεύουμε ότι η κοινωνική νομολογία, θα πρέπει, νομοθεσία θα πρέπει να είναι σαφής. Ένα νέο σενάριο της εσωτερικοποίησης του κόστους θα πρέπει να είναι σαφές και να γνωρίζουμε μέχρι πού θα φτάνει η νομοθεσία των κρατών μελών και μέχρι πού θα πηγαίνει η νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το τελευταίο θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα και με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετα, μετατραπεί σε έναν εγγυητή δημόσιο σε θέματα ασφάλειας όσο και αηφορίας του κλάδου. Αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν χρειάζονται προσαρμογές στον προϋπολογισμό και η Επιτροπή μας ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να παράσχει μηχανία να ανακαλύψει η βιομηχανία ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των δαπανών. Πιστεύουμε ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν θα πρέπει να εξαρτώνται άμεσα από τις διακοιμάσεις των αγορών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και η διασύνδεση με τον συγκεκριμένο κλάδο. Έχουμε προτείνει λοιπόν ως του ένα σταθμισμένο σύστημα χρηματοδότησης όπου καταβολές από πλευράς επιχειρήσεων είτε πρόκειται για τέλος είτε για άλλο τρόπο, είτε για άλλο τρόπο θα πρέπει να λειτουργεί πάντα σε σχέση με την ε, βιωσιμότητα του κλάδου αλλά και το του και πρωτίστως της ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους ε, ε, αυτή είναι μια πρόταση που έχουμε καταθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει να πάρει κάποιο το λόγο. Κύριε Καλβίνιο, θέλετε να λάβει το λόγο. Όχι, η Κομισιόν δεν επιθυμεί να μιλήσει. Δεν το επιθυμεί. Α, το επιθυμεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Μια κάποια αντίδραση σε σχέση με τα σημεία τα οποία θίγησαν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το σύστημα χρηματοδότησης που ισχύει, που είναι ένα υβριδικό σύστημα, με τα τέλη, με τα κονδύλια τα οποία ανταποκρίνονται στα, στα τέλη των επιχειρήσεων. Αυτό το πρότυπο λοιπόν έχει μια κάποια περιπλοκότητα, αλλά δεν οδήγησε σε δυσκολίες χρηματοδότησης. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν υπήρξε ανεπάρκεια χρηματοδότησης ε, για την υπηρεσία. Σχετικά τώρα με το να μεταβούμε σε ένα σύστημα που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη βιομηχανία, ε, κίνδυνοι αναφέρθηκαν από πολλούς παρεμβαίνοντες και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξάρτηση της υπηρεσία και τις ειδικέ υπηρεσίε που αφορούν στις βιομηχανίες. Επίσης, σε περίπτωση που όλα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τέλη που θα καταβάλει η βιομηχανία, ο κίνδυνος ε, του να υπάρξει κάποια σύγκρουση συμφερόντων και μια ανισορροπία του τομέα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το παράδειγμα των υπηρεσιών που γνωριδοτούνται κατά 100% από τα τέλη της βιομηχανίας που στο παρελθόν ε, οδήγησαν σε πλεονάσματα τα οποία είχαν ε, επιπτώσεις ε, όπως ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εθνικών Υπηρεσιών εκπροσωπούνται και όπου η συμμετοχή της Ένωσης είναι κάπως απομακρυσμένη θα λέγαμε, έχει διακόψει κάπως ε, την συνέχεια και έχει υποβάλει τη βιομηχανία σε περισσότερα έξοδα από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα, για το θέμα της χρηματοδότησης επίσης, να πω ότι στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ε, των υπηρεσιών υπάρχει η Επιτροπή, η Ομάδα Εργασίας που προβλέπεται τον Οκτώβριο να εξετάσει τα πρότυπα χρηματοδότησης ε, μέσω άλλων ε, οδών πέραν του προϋπολογισμού της Ένωσης και να μπορέσει να εξετάσει τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Γκάγερ στο στην έκθεσή του και να καθορίσει ένα δόγμα μακροπρόθεσμο θα έλεγα, όχι για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στην βιομηχανία, στον κλάδο δηλαδή. Πιστεύω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι υπηρεσίες ε, δεν έχουν έφεση να διαπιστώνουν πλεονάσματα και ωφέλη, κέρδη. Και συνήθως θα πρέπει να τιμολογούν ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία. Αν υπάρχει πλεόνασμα σε κάποια υπηρεσία, αυτό σίγουρα μπορεί να σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές φοβόντουσαν ότι θα υπήρχε ανταγωνισμός και ότι υπήρξε υπερτιμολόγηση, κάτι το οποίο σίγουρα οδήγησε σε συσσόρευση ε, ποσών, ε, εξού και πλεόνασμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να ελέγξουμε τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αυτές υπηρεσίες. Ο εισηγητής κ. Γκάιερ, ε, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. πώς να το πω, μελέτησα την ιδέα για κάποιο διάστημα, α το πω ίσω κάπως υπερβολικά, να είναι πλήρως ιδιωτικός χρηματοδοτούμενοι πολλοί οργανισμοί. Πολλοί οργανισμοί, περισσότεροι από Και για εκείνους όπου είχαμε εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πολλοί με θεωρούν ύποπτο μια τέτοιας πρόθεσης. Αλλά δεν το έχω γράψει το κείμενό μου πάντως αυτό. Εάν κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλεί παρανοήσεις, ευχαρίστως να επανεπεξεργαστώ το κείμενο και να συνεργαστώ μαζί σας για να φτάσουμε σε ξεκάθαρες διατυπώσεις. Και για να το πω με απόλυτη σαφήνεια, δεν έχω ενδιαφέρον ως εισηγητής να κάνω τον ΕΑΣΑ πλήρως ιδιωτικός, δηλαδή από τα τέλη, τις φορές των επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμενο οργανισμό. Διότι πολλά από τα επιχειρήματα των συναδέλφων είναι σωστά και με βρίσκουν σύμφωνο. Εάν για να υπάρξει αυτή η σαφήνεια πρέπει να ξανακοιτάξουμε το κείμενο, ευχαρίστως να το ξαναδώ όχι μόνο με τους σκιώδεις και εισηγήτριες, αλλά όποιος επιθυμεί να συμβάλλει στην διευκρίνηση, ευχαρίστω. Αυτό που εννοώ με τα όσα είπα πριν είναι ότι αυτή η μέχρι την τελευταία δεκάρα διάκριση των δύο ειδών καθηκόντων του ΕΑΣΑ πρέπει να διευκολυνθεί με την έννοια ότι τα τέλη που καταβάλει βιομηχανία και σωστά είπε η κυρία Χολμάιρ δεν μπορούν να μετρώνται μόνο στη βάση του πραγματικού κόστους αλλά στην βάση εκτιμήσεων εάν ακολουθήσουμε άλλο σύστημα χρηματοδότησης Τι κερδίζουμε. Ας το πω ξανά λοιπόν. Δεν με ενδιαφέρει ένας οργανισμός που να είναι πλήρως ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος κατά 100% και που εν τέλει ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων κόστους της ΕΑΣΑ θα αναλαμβάνεται από τον δημόσιο προϋπολογισμό. Αυτό πρέπει να διευκολυνθεί, αυτό εννοώ. Ούτε είναι επιθυμία μου να επιβάλλουμε υπερβολικά υψηλά τέλη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διότι η ΆΣΑ προσφέρει και υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα και αυτού του είδους οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται από δημόσιους προπολογισμού. Αυτό που με δυσκολεύει είναι ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση να μειωθεί κατά 5% ο αριθμός των εργαζομένων. Μπορώ να το δεχτώ γενικότερα για τις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά εδώ πρόκειται για φορέα παροχής υπηρεσιών. Περί αυτού πρόκειται. Και δεν μπορούμε, παραδείγματο χάρη, σε ένα τομέα όπως τις ε, αερομεταφορές, την πολιτική αεροπορία, αλλά και έναν οργανισμό που αφορά μια ρυθμιστική αρχή. Η δαπάνη σε αυτούς τους ε, οργανισμούς καλύπτεται από την αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το θέμα είναι να μην υπάρχει να μην υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ αυτών που ζητούν παραδείγματο χάρη μια πιστοποίηση και αυτών που καταβάλουν τα κονδύλια, που χρηματοδοτούν. Οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν πριν τις 25 Μαΐου στις 10 το πρωί. Η οθέτηση Αρχικά είχε προβληθεί για τις 30 Ιουνίου. Καταλαβαίνετε όμως ότι η 30 Ιουνίου είναι μετά τις 23 Ιουνίου και εκεί θα έχουμε πληθώρα θεμάτων. Άρα η έκθεση του κυρίου Γκάγερ θα πρέπει να υιοθετηθεί στις 27 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Επιτροπή Τρανς θα ψηφιστεί και στην Ολομέλεια κάποια στιγμή το φθινόπωρο, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γκάιερ. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι η μέσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Θα δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές και δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο πρώτος, η κυρία Τομά ή ο κύριος Όλμπριτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς καταρχήν γιατί δεχτήκατε να αναβάλουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε, εγώ δεν το έκανα πολύ εύκολα αυτό, καθότι δεν μου αρέσει αυτό που έχουμε αποφασίσει να μην αναπνέουμε, δηλαδή να μην κάνουμε τίποτα μέχρι τις 23 Ιουνίου, σαν να υπάρχει ένα εθνικό θέμα το οποίο υπερέχει των ευρωπαϊκών. Κοιτάξτε, και εμένα μου στήχησε και βεβαίως ε, εδώ προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε κάποιους Βρετανούς συναδέλφους. Από την άλλη, το ότι ψηφίζουμε την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πολιτικού ε, πλαισίου τέσσερις ημέρες μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα θα δώσει στην ψηφοφορία αυτή έναν επίσημο χαρακτήρα, τον οποίο πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικό. Έκθεση λοιπόν του κυρίου Γκάγερ και η δική μου θα είναι οι πρώτε ψηφοφορίε που θα λάβουν χώρα μετά το Βρετανικό ε, δημοψήφισμα και βεβαίως ε, του δίνει και μια βαρύτητα. Εάν ήσασταν ε, Βρετανοί υπήκο, τι θα λέγατε, κάτι μας κρύβουν. Όχι, αφού πρόκειται για δημόσιο έγγραφο το συζητούμε, αλλά εν πάση είναι δημόσιο έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλες τις πολιτικές ομάδες, όλους τους συναδέλφους για τις 328 τροπολογίες που υποβάλλατε. Έχουμε εξετάσει κάποιες από αυτές ήδη και νομίζω ότι σήμερα Οι συνάδελφοι με πάθος ε, θα παρουσιάσουν ε, τις τροπολογίες αυτές, θα τις υποστηρίξουν. Οι περισσότερες από αυτές εξάλλου, και εγώ και ο κύριος Όλμπριχ τις δεχόμαστε με χαρά, καθότι πάνε προς την σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικοδομητικό για την ε, εργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. Πρέπει να δείξουμε πνεύμα συνένεσης και σίγουρα οι τροπολογίες σας εμπλουτίζουν το αρχικό μας κείμενο. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι με τον συνάδελφο, τον Γιάνν Όλμπριχτ, συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τροπολογίες, κάποιες από τις τροπολογίες, οι οποίες είναι κάπως εκτός θέματος. Ό,τι έχει σχέση, παραδείγματο χάρη, με την μακροοικονομία, ό,τι έχει σχέση με την ζώνη ευρώ, ό,τι έχει σχέση με την αιρεσιμότητα, με μακροοικονομικούς ε, στόχους. Πρόκειται για αρμοδιότητες άλλων επιτροπών. Παραδείγματο χάρη, αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής όλοι όσοι υπέβαλαν τέτοιες τροπολογίες από την αρχή του 2017 θα αρχίσει η συζήτηση αυτή και εκεί μπορείτε να υποβάλλετε ό,τι τροπολογία θέλετε για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σήμερα όμως το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει και δεν μπορεί να ενσωματώσει τέτοιες τροπολογίες. Το ίδιο θα έλεγα και για τη συνοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν να ενσωματώσουμε τροπολογίες που δεν εμπίπτουν στο θέμα μας. Για όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες και ο Γιάνν Όλμπρεχτ και εγώ θέλουμε να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε τροπολογίες οι οποίες έχουν σαν σκοπό να εξαλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δηλαδή σκοπός μας είναι να μειώσουμε, να μειώσουμε, να μειώσουμε την εμβέλεια της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής και της χρηματοδότησης από τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ε, όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, πρέπει να είμαστε, επαναλαμβάνω, ανοιχτοί να δείξουμε πνεύμα συνένεσης και θα το κάνουμε και ελπίζω στις 27 Ιουνίου να είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο τέσσερις μέρες μετά το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τόμα. Ο κύριος Όλμπρεχτ. Να, προσφέρω, να προσθέσω κάτι. Προς το παρόν έχουμε 358 τροπολογίες αλλά έχουμε μόνο δύο γνωμοδοτήσεις ε, από την Εξειδικευμένη Επιτροπή. Περιμένουμε τις υπόλοιπες γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών. Ε, περιμένουμε να βρούμε χρόνο για να δουλέψουμε πάνω στις τροπολογίες και επί των συμβιβασμών που θα καταστούν δυνατοί, αλλά πιστεύω πως ε, σήμερα είναι μάλλον τα μέλη της Επιτροπής μας που έχουν παρουσιάσει τις παρατηρήσεις τους δεν πρέπει να επαναλάβουμε σήμερα αυτά που έχουμε ήδη ξαναπεί στο παρελθόν. Πιστεύω ότι να συμφωνήσουμε με κυρία Τομάς ότι ίσως τώρα η συζήτηση επί του προϋπολογισμού περισσότερο από ποτέ αντανακλά την συζήτηση επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για μια τεχνική συζήτηση είναι πολιτική η συζήτηση στην ουσία. Λοιπόν, στη συζήτησή μας και στις ψηφοφορίες που θα διεξαχθούν θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη ανάμεσα στα μέλη που θα παρουσιάζουν την φιλοευρωπαϊκή στάση τους, αλλά από την άλλη πλευρά θα υπάρξουν μέλη τα οποία δεν ε, είναι ε, είναι μάλλον πολέμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μπαίνουμε στην πολιτική ζήτηση και για να κλείσω αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τη ζήτηση. Μετά θα ακούσουμε την Κομισιόν. Δεν πρέπει να παραμείνουμε παθητικοί. Χρειάζεται να γνωρίζουμε την άποψη της Επιτροπής αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι θα είμαστε ενεργοί σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου που θα συζητεί το θέμα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από το δημοψήφισμα το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι θετικό για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρώτα να δώσω το λόγο στους πιο και ευχαριστώ για μια ακόμα φορά τους δύο συνεισηγητές κυρία Τωμά μας είπε ότι υπάρχουν τροπολογίες ε, που μπορούν να γίνουν δεκτές, άλλες ε, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτες, αλλά υπάρχει και το ζήτημα της γεωργικής πολιτικής, ε, το οποίο δεν συζητείται εδώ. Υπάρχουν και κάποιες αμφισβητήσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε υπολογίσει τον αριθμό των τροπολογιών από τις 358 δηλαδή, ποιες είναι οι παραδεκτές και μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες συμβαστικές προτάσεις χωρίς μικρόφωνο. Πιστεύω πως το μεγαλύτερο τμήμα των τροπολογιών αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δημοσιονομικό Δύσκολα θα συντάξουμε σήμερα ε, συμβασμούς, αλλά Ακούγοντας τους σκιώδεις ηγητές θα δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Κολμέν μπορεί να μας πει τη γνώμη της πολιτικής ομάδας. Ομολογώ κύριε Πρόεδρε ότι η ενημέρωση που διαθέτω δεν μου επιτρέπει να συμβάλλω ουσιαστικά στην ε, συζήτηση. Ε, λυπούμε λοιπόν και ε, προτιμώ να μην συμμετάσχω. Εάν ήταν ανάμεσα μας και ο Ντεπρέ θα είχε σίγουρα εκφραστεί. Ή ο κύριος Τόρβαλτς αν ήταν παρόν αυτός, αλλά ούτε και αυτός είναι. Η κυρία Νίριάντα. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Οποιουσδήποτε θα υπέφερε από πονοκέφαλο με τόσες πολλές τροπολογίες. Τους ευχαριστώ λοιπόν που έκαναν την δουλειά αυτή. μα ενδιαφέρει και μας ο εν ώψη και του ενδεχόμενου Brexit. Οφείλουμε να εξετάσουμε προσεκτικά το ενδεχόμενο αύξηση των οροφών. Μιλούμε για αυτά. Είναι μέγα το θέμα. Χρειάζεται κάποια ρεαλιστική προσέγγιση για το πώ θα το κάνουμε και επίση η αύξηση των ενισχύσεων, των στήριξεων που δίνουμε για ε, πρόσφυγες και μετανάστες και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά βέβαια συναποτελούν ένα ε, σύνολο. Ελπίζω και εύχομαι η συζήτηση να συνεχιστεί. δίκα τα λόγια ο κ. Μαραγκάλ. Εκτός μικροφώνου. Να ευχαριστήσω τους συγητές για το έργο τους Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ καλό πλαίσιο εργασιών. Να πω επίση ότι θα το ψηφίσουμε φυσικά σήμερα, αλλά είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε τον χρόνο για να το ψηφίσουμε και να πω ότι αυτή πρέπει να είναι η έκθεση αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον γλώσσο και την ορολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις δηλώσεις του Ευρωκοινοβουλίου και με την πεποίθηση, με κάποια αισιοδοξία και με υπερηφάνεια. Είναι ένας προεκλογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι προεκλογισμός ε, μιας ε, επιμέρους χώρας. Έχουμε υποβάλει 70 τροπολογίες. Πολλές ακούγονται, φυσικά κάποιες από αυτές ε, θα θα μειωθούν, αλλά 10-12 νομίζω θα είναι αυτές που ε, θα ε, περιλάβουν το, τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Υπάρχουν θέματα ποσοτικά και ποιοτικά. Τώρα από ποσοτικά επανειλημμένα αναφέρουμε την Αγία για αύξηση των ορίων των ανωτάτων ορίων, αλλά δεν θέτουμε ούτε κριτήρια, ούτε ποσότητες, ούτε κάποια κατά προσέγγιση ποσά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο όριο το 1,29% θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 150 εκατομμύρια ανά περίοδο. Δεν είναι πολλά, είναι αρκετά αλλά όχι πολλά. Το χαμηλότερο κατώτερο όριο θα πρέπει να είναι η πρόταση της Κομισιόν και γι' αυτό υφίσταται 85 δις. Αυτά είναι τα όρια που θα πρέπει να μας... Ε, σε αυτά τα όρια θα πρέπει να παραμείνουμε. Τέλος θα έχουμε την ευκαιρία για να το πράξουμε. Τώρα, από πλευρά ποιοτική, νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία για να προσδιορίσουμε ένα πλαίσιο για αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές σύμφωνα με τις πολιτικές που έχουμε αποφασίσει. Ό,τι αποφασίζουμε σήμερα θα πρέπει να προσανατολίζεται ε, στα θέματα της πολιτικής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 με τους συγκεκριμένους στόχους τους των περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς. Έχουμε στόχους λοιπόν, έχουμε targets. Ε, το πώς θα τους πετύχουμε. Άλλο κριτήριο θα πρέπει να είναι η εσωτερικοποίηση των διεθνών μας υποχρεώσεων. Νομίζω ότι Οι κραυγές που ακούγονται σήμερα είναι αυτές που προέρχονται από τα άτομα τα οποία απομακρύνονται σήμερα από την ειδωμένη. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ε, ακούμε σήμερα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, στόχοι μεσοπρόθεσμοι, μεσομακροπρόθεσμοι κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να κοφεύουμε σε αυτές τις κραυγές που ακούγονται σήμερα. Πρέπει επίση να βρούμε μια καλύτερη συνέργεια ανάμεσα στην ε, ανταγωνιστικότητα και την συνοχή. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια με τη στρατηγική 2020 και τέλος Πρόεδρε, για μετά το 2020, δύο πράγματα δεν ναι, βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να αφισβητήσουμε αυτή την προοπτική που αφορά το μετά 2020. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετική με τους πόρους. Ξέρουμε ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να ζητηθεί στο High Level Group, το οποίο δεν ε, έχει δημιουργηθεί ακόμα, δεν έχει συσταθεί. Και φυσικά δεν θα πρέπει να αποκλείουμε νέες ιδέες, ε, νέες έννοιες, ε, όπως τα Financial ε, Transaction Tax και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίζουν, προβληματίσουν από τώρα που αφορούν το μετα, περίοδο μετά το 2020. Χρειάζεται λοιπόν να υποστηρίξουμε έναν προπολογισμό ο οποίος θα είναι ελεύθερος από δεσμεύσεις διμέρεως ε, περιεχομένου. Ευχαριστώ. Με εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ κύριο Ζαντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τους δύο εισηγητές για το έργο τους και τους εύχομαι καλή επιτυχία και καλό κουράγιο για την ανάλυση αυτών των τροπολογιών. Τώρα, η θέση μας ε, η οποία ε, αντικατοπίζει τις θέσεις που έχουμε συμπεριλάβει στις τροπολογίες μας είναι μια θέση, μια στάση η οποία προσπάθησε να συμπεριλάβει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά αυτής της έκθεσης που είναι περισσότερο πολιτικής φύσης αλλά που φτάνει σε μια δύσκολη κατάσταση το ιστορικό της Ένωσης. Όπως είπαν οι προελίσσαντες, σε αυτό το ζήτημα, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ρεαλιστικοί. Πρώτον, να πούμε ότι ενωσιακό προπολογισμό δεν μπορεί αλλά και ούτε πρέπει να επιλύει όλα τα προβλήματα της Ένωσης. Κάθε τόσο και πολύ συχνά ζητάμε περισσότερα από το, σε δυνατότητες αυτού του προπολογισμού και οι δυσκολίες φυσικά είναι προφανείς κατά την διαχείριση αυτών των λίγων πόρων. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μια οικονομική κατάσταση απόλυτα ασταθή και κάποιες φορές καταστροφική. Να κάνουμε λοιπόν μια εργασία ορθολογικοποίησης των δαπανών. Πρέπει να, είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να κατανοήσουμε ποια προγράμματα, ποιες δαπάνες είναι πράγματι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν με τρόπο αποτελεσματικότερο και ε, σε εθνικό επίπεδο και ποιες σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάποια μακροπρογράμματα σήμερα αυτό το θέμα θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ε, επί των ίδιων αυτών ζητημάτων και εργαλείων που έχουμε συστήσει το τελευταίο καιρό για την εντοπίση το προβλημάτων που έχει γνωρίσει η Ένωση, παραδείγματο χάρη η κρίση των μεταναστών, το προσφυγικό ζήτημα, η κρίση του θέμα των επενδύσεων, υπάρχουν και το πρόγραμμα Juncker, όπου έχουν χορηγηθεί, προβλεφθεί μάλλον να χορηγηθούν τεράστια ποσά και με την πρώτη έκθεση που έχει συντάξει η Κομισιόν βλέπουμε τα αποτελέσματα τα οποία είναι απόλυτα ε, μη ικανοποιητικά. Δεύτερον, η συμφωνία με την Τουρκία. Δισεκατομμύρια ευρώ βγαίνουν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και βλέπουμε ότι με τα δυσκολία εφαρμόζεται η εν λόγω συμφωνία. Και νομίζω ότι Αυτά τα οποία λαμβάνει η Ένωση από τη συμφωνία αυτή από την με την Τουρκία δεν ε, είναι αρκετά και δεν είναι διόλου Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα εξετάσουμε διάρκεια των συζητήσεων και συναντήσεων που θα έχουμε με τους συγητές, με τους, με τους ε, σκιώδεις Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζουλτέκ δεν είναι εδώ. Και τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Να, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σοσιαλιστική ομάδα συνέβαλε και αυτή με κάποιες τροπολογίες. Ελπίζουμε πως οι συγητές δεν θα μας κάνουν μούτρα επειδή προσθέσουμε δουλειά στο ε, έργο τους. Φυσικά θεωρούμε ότι αυτές οι τροπολογίες ε, δεν ε, είναι αντίθετες με το έργο των δύο συνεισηγητών, απλά θελήσαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα κάποιες πτυχές. Δεν θα επισέλθω σε όλες, αλλά σε αυτές που για τους σοσιαλιστές είναι σημαντικότερες. Πρώτον ότι έχει σχέση με τους ιδίους πόρους, μιλάμε για τις ταπάνες και εδώ θα δαπανηθούν ε, κονδύλια από το δημοσιονομικό πλαίσιο, το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερους πόρους και ως εκ τούτου απαιτείται να δευκνήσουμε καλύτερα τις ε, φόρους και τα τέλη τα οποία συζητώνται και αν θα μπορέσουμε να ε, απαλύνουμε τον ε, πληρωμές που καταβάλουν τα κράτη-μέλη. Το καταπολέμηση επίσης της φοροδιαφυγής. να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εργαστεί για ένα αρμονισμένο φόρο εταιριών. Υπάρχει ένα δεύτερο, μια δεύτερη δέσμη τροπολογιών που έχουν σχέση με την COP21, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το ε, θέμα της βιοπικιλότητας ε, που δεν υπήρχε ακόμα στο τραπέζι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου ε, είναι απαραίτητη. Μια τροπολογία που έχουμε καταθέσει που αφορά την ΚΑΠ για να, να αποφυγεί η χρηματοδότηση νέων πολιτικών ήδη κατεβλήθη προσπάθεια στο παρελθόν μείωση των κονδυλίων που δαπανούνται για αυτή την πολιτική, αλλά θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει ένα τμήμα αυτών των κονδυλίων να δοθεί για χρηματοδότηση νέων πολιτικών για του πρόσφυγε. Θέλετε να τονίσουμε την ε, ευθύνη των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας και ξεπερνάνε κατά κάποια δέκατα των, ε, τις υποχρεώσεις θεωρούμε ε, ε, τους επιβάλλουμε κυρώσεις. Θα πρέπει λοιπόν και τώρα να επιβάλλουν κυρώσεις εάν οι χώρες δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των μεταναστευτικών και των προσφυγικών. Το ζήτημα τώρα του αποθέματος για αντιμετώπιση κάποιων κρίσεων θα πρέπει να υπάρξει ένα αποθεματικό για αντιμετώπιση κρίσεων της τάξης του 1,23. Τέλος, η, σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη συζήτηση και τις τροπολογίες των Βουλών 2017 και το δημοσιονομικό πλαίσιο και η αναθεώρηση αυτού. Όχι για ζήτημα στρατηγικής, ούτε για θέμα άσκησης πίεσης ή απειλών. Είναι ζήτημα λογική. το μιλάμε για αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου που θα πρέπει να επηρεάσει το προπολογισμό 2017 μέχρι το 2020, δεν θα ήταν λογικό να διαπραγματευτούμε έναν προπολογισμό για το 2017 δίχω να λαμβάνουμε υπόψη το δημοσιονομικό πλαίσιο και πώς αυτό θα επηρεάσει τον προπολογισμό. Αυτό λοιπόν εν γέννη και οι κατευθύνσεις γραμμέ που μα καθοδήγησαν. Ευχαριστώ. κύριος Ντεσόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω σύντομα. για, την, ε, για λογαριασμό της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπου είμαι σκιώδης συγητής και όπου είναι πολύ επικοδομητική η ατμόσφαιρα. Δεν προτείνουμε τροπολογίες, Είμαστε κατά αυτής της στάσης που πάει να καταστρέψει τον προπολογισμό για πολλά σημαντικά πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό για το Λαϊκό Κόμμα και είναι σημαντικό να δοθεί το μήνυμα στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα εν προκειμένου. Το ένα είναι οι μεταναστευτικές ροές και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν αλλάξει τις πολιτικές προτεραιότητες στην Ευρώπη και για το λόγο αυτό είναι κρίσιμο να επανεξεταστεί το ΠΔΠ. Η θέση μας επίσης είναι, ε, περιλαμβάνεται σε 36 τροπολογίες, με πέντε πολύ ε, θετικές συμβαστικές τροπολογίες. Ψηφίζουμε την επόμενη εβδομάδα εμείς και νομίζω ότι θα προτείνουμε κάποιες λύσεις σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ Γιάν και ευχαριστώ και εσάς Ιζαμπέλ για την θαυμάσια δουλειά που έχετε κάνει. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Μάνκα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ και τους δύο συγκητές για την δουλειά που έκαναν. Ερώτηση προς την Κομισιόν. ζητήσαμε από την Κομισιόν να συντάξει μελέτη αντικτύπου στην βάση της οποίας να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις για τις περαιτέρω φάσεις του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου γιατί υπάρχουν και καθυστερούμενες πληρωμές και μέσα στον τριμηρή διάλογο αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτη αντικτύπου για τον αντίκτυπο ακριβώς των καθυστερουμένων πληρωμών μέχρι το 2015. Για τις επιπτώσεις δηλαδή των καθυστερήσεων αυτών πληρωμών στο σύνολο της εκτελέσεως του προϋπολογισμού και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα άλλο πράγμα που ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει είναι η στήριξη της απασχόλησης των νέων. Ίσως να ενθυμίσετε στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις είχαμε συμφωνήσει ότι θα ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να μας δώσουν μια συνολική αξιολόγηση, από την Επιτροπή μάλλον, μια συνολική αξιολόγηση για τις επιπτώσεις της πολιτικής στήριξης της απασχόλησης των νέων στις διάφορες χώρες μέλη. Και έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε ζητήσει μέχρι τέλη του Απριλίου 2016 να μας υποβάλει σχετική μελέτη αντικτύπου επιπτώσεων. Δεν την έχω δει όμως εγώ ακόμη, δεν ξέρω αν έχει υποβληθεί καν. Το τρίτο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γνωρίζουμε ότι το Ταμείο αυτό υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτεί επενδύσει υψηλού ρίσκου που δεν θα ήταν δυνατό να αναλυθούν χωρίς το Ταμείο αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν έργα, για παράδειγμα ένα για την θέρμανση 40.000 διαμερισμάτων. το οποίο θα μπορούσε να γίνει και χωρίς την παρέμβαση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αλλά θα έπρεπε να είχαμε κόψει άλλα πράγματα. Όντως λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις αυτές δίνονται μόνο σε έργα υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Χρειαζόμαστε τις προφορίες αυτές για να μπορέσουμε να λάβουμε περαιτέρω αποφάσεις αν δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά, δεν μπορούμε να λάβουμε τι αποφάσει αυτέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν τι μελέτε αντικτύπου. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς κύριε Νεγκρέσκου. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ του δύο εισηγητέ. Θέλω όμω να υπογραμμίσω κάτι όσον αφορά τη διατύπωση κάποιων άρθρων είναι σαν να ζητάμε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική συνοχής, στα ταμεία συνοχής. Εγώ θεωρώ ότι αν ε, ζητήσουμε κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Αν αρχίσουμε δηλαδή τώρα μια μεγάλη συζήτηση για την αναδιάρθρωση των ε, ταμείων συνοχής, αυτό δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Οι χώρες που σήμερα προσπαθούν να καλύψουν την διαφορά ανάπτυξης, οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, χρειάζονται αυτή την πολιτική. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε περισσότερη αλληλεγγύη και να αρχίσουμε και επικρίνουμε τα ταμεία συνοχής. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η πολιτική αλληλεγγύης για αυτές τις χώρες κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί. Είναι κάτι που το διαστανόμαστε, είναι κάτι που έχει γίνει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά αυτό που ζητάμε και από τα κρατημέλη αλλά και από την ε, Επιτροπή, αυτά αποτελέσματα δηλαδή, ιδιαίτερα για τα προγράμματα αυτά τα οποία ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους νέους, όχι μόνο αυτοί που βρίσκονται σήμερα εκτός αγοράς εργασίας, αλλά και για όλους τους νέους. Ενδεχομένως να πρέπει να ενισχύσουμε λίγο παραπάνω την πτυχή αυτή ε, των προτάσεων που αφορά τους νέους. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στους και στην Επιτροπή. Κάτι που δεν μπορεί να ενσωματωθεί τώρα σε τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι προτείνει ένα είδος σχέδιο που αφορά την Αφρική. Που βασίζεται σε ένα μοντέλο χρηματοδότησης ταμείου για να φτάσουμε σε ένα συνολικό ποσό χρηματοδότησης 60 δισεκατομμύρια έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές από κάποιες χώρες της Αφρικής από τις οποίες φεύγουν οι περισσότεροι. Ένα είδος συμφωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης με τις χώρες αυτές για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των ροών, των μεταναστευτικών ροών. Ένα είδος ταμείου συνεργασίας και ανάπτυξης για την Αφρική. Έχουμε αναβάλει τη συζήτηση βεβαίως. Θα μπορούσαμε όμως εντωμεταξύ να επεξεργαστούμε και αυτή την πρόταση, καθότι σίγουρα θα έχει επιπτώσεις επί της αναθεώρησης. Αν δηλαδή υποβληθεί μια τέτοια πρόταση από την Επιτροπή, σίγουρα αυτό θα συμπεριληφθεί στην αναθεώρηση. Εγώ προσωπικά άκουσα αυτή την ιδέα, την βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Το διάβασα στον τύπο βέβαια, δεν ξέρω ακριβώς ε, περί τίνος πρόκειται. Αλλά οι δύο συγητές θα μπορούσαν μέσω πρότασης τροπολογίας ε, των εισηγητών να συμπεριλάβουν αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας δώσει περισσότερες διευκρινήσεις η Επιτροπή όταν πάρει το λόγο. Θα μας πει αν προετοιμάζεται κάτι τέτοιο και αν μπορεί αυτό να συμπεριληφθεί πριν από τις 23 Ιουνίου, κ. Μπέγκε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δύο για το έγγραφο. Για τις κατηγορίες 3 και 4 έχω καταθέσει τροπολογίες. Ωστόσο, μια παρατήρηση για τα όσα είπε ο κ. Νεγκρέσκου προηγουμένω. Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί μονόδρομο. Τα διαρθρωτικά ταμεία δημιουργήθηκαν κάποτε με συγκεκριμένο σκοπό. Είναι θεμητό λοιπόν από τη μια μεριά να ζητούμε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις όλων. Δηλαδή να μην αγγίξουν τους εθνικούς φακέλους, envelopes δηλαδή, στα πλαίσια της αναθεώρησης. Το εάν τώρα πρέπει να επαγγελματοποιηθούν περαιτέρω τα ταμεία για να στηρίξουν περισσότερο την απασχόληση, αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό καθήκον το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θέλω επίσης να επανέλθω στα όσα μόλις είπε η κυρία Μπρέσο σήμερα το πρωί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προπολογισμών μίλησα και συνέδεσα ορισμένες ερωτήσεις με το θέμα αυτό, διότι τίθεται το ερώτημα, όντως, εάν τα όσα ακούγονται τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέπτεται να καταθέσει πρόταση αρχές Ιουνίου της τάξης των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό στα πλαίσια του ΕΦΣΙ και στα πλαίσια των ε, χρηματοδοτήσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για το Κοινοβούλιο, θα θυμόμαστε όλοι την εποχή όπου γινόντουσαν οι συζητήσεις για το ΕΦΣΙ και όπου είχαν παραμερίσει κάποιες επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου. Θα θυμούμεθα όλοι, θα όλοι και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί τότε για να διορθωθεί η πορεία. Προφανώς συζητείτε για κάτι που θεωρώ σωστό. Εφόσον δηλαδή κάποια κονδύλια γίνονται decommitted, δηλαδή φεύγουν από τον προϋπολογισμό, χάνονται για τον προϋπολογισμό, να χρησιμοποιηθεί ευκαιρία για να γίνουν κάποιες μετακινήσεις πιστώσεων και να προκύψουν κάποιες, κάποια νέα καθήκοντα για τις πιστώσεις αυτές. Είμαι υπέρ και αυτή τη ιδέα. Νομίζω όμω και ενδεχομένω η Γενική Διευθύντρια τη Κομισιόν να μπορέσει να μα βοηθήσει εν προκειμένου Νομίζω ότι αυτό δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στο να γίνει πρόταση, όπως έχει ανακοινωθεί, με την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων θα έρθει στις 28 Ιουνίου να εγκρίνει το σχετικό πακέτο. Διότι δεν έχει τέτοια νομοθετική αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι, τότε το Κοινοβούλιο κάποια στιγμή πρέπει να στραφεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και το άλλο θέμα, κυρία Γενική Διευθύντρια, είναι η προσέγγιση για την αναθεώρηση. Δεν νομίζω ότι αρκεί. Διότι ναι μεν οι σκέψεις είναι σκόπιμες που έχουν γίνει σχετικά με το μέγεθος των κονδυλίων για τη σταθεροποίηση των γειτονικών με την Ένωση χωρών, αλλά σημαντική είναι επίσης και η ποιότητα των προγράμματων, ώστε να επιτύχουμε περισσότερα θετικά πράγματα από ό,τι έχουμε επιτύχει προφανώς μέχρι τώρα, το πρόσφατο παρελθόν δηλαδή. Ταυτόχρονα όμως, σήμερα, τις μέρες αυτές τουλάχιστον, σε συνάντηση, σε συνάντηση κορυφής που διεξάγεται στην Τουρκία με συμμετοχή δεν ξέρω πόσων χωρών μελών, συζητούνται οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και τα Ηνωμένα Έθνη και βλέπουμε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στο παρελθόν να μην υλοποιούνται. Στα πλαίσια της αναθεώρησης της δημοσιονομικής προοπτικής και των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ή άλλως είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές, πρέπει να σκεφτούμε και μια μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση, για παράδειγμα, του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για αντιμετώπιση μεταναστευτικών και προσφυγικών θεμάτων κλπ. Που εξαντλήθηκε το 2014. Και ποιο είναι το συμπέρασμα που συνάγουμε από το γεγονός αυτό για τον χρηματοδοτικό σχεδιασμό. Και το πολύ σημαντικό θέμα έγινε ένας αναπρογραμματισμός που απίτησε σημαντικότατη δημιουργικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που για να μπορέσουν να απαντηθούν αυτά, μπορεί να απαντηθούν αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις μέχρι το 2020. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε με το πρόβλημα των πληρωμών, διότι αυτές παραμένουν εκκρεμείς. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει μεγάλη ευθύνη. Την μεγάλη ευθύνη να τα συνδυάσει σωστά όλα αυτά τα πράγματα και να δώσει ξεκάθαρο μήνυμα ως το θεσμικό εκείνο όργανο το οποίο διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό στον τομέα αυτόν. Είτε δηλαδή θα επιλέξουμε μια σωστή προσέγγιση την οποία θα διαπραγματευτούμε μετά είτε θα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας όπου εν τέλει όλα θα καταρρεύσουν. Αυτά πρέπει να συζητηθούν και στις αρχές των διαπραγματεύσεων, αλλά και στην τελική επεξεργασία του κειμένου. Και μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια. Ευχαριστώ. Ο κ. Σάββαμα, τελευταίος παρεμβαίνουν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, το θαυμασμό μου θα έλεγα, προς τους δύο εισηγητές, έχετε δίκιο. Πρόκειται περί θαυμασμού ουσιαστικά. Πραγματικά. Και λίγα λέω. Ουσιαστικά εδώ πρόκειται για μία πολύ γερή δομή και πραγματικά δεν θα συνεχίσω λέγοντας πόσο καλή είναι η εργασία σας. Ε, θα περιοριστώ μόνο σε κάποια πράγματα που με ανησυχούν σε αυτήν την πολύ θωρακισμένη δομή. Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στον κατεπήγοντα χαρακτήρα κάποιων διαδικασιών. Ο κύριος Μπέγκε το ανέφερε. Τα επόμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν τα επίγοντα θέματα θα πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί εδώ ακούμε τι συνέβαινε στο παρελθόν και τι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σήμερα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω τώρα να τα αμφισβητήσω όλο, όμως ε, σίγουρα και σε θέματα ε, γεωργίας και στην παράγραφο 20 που αναφέρονται τα πολιτιστικά. Σε καμία περίπτωση ε, αυτό δεν είναι αντιφατικό με την κοινή αγροτική πολιτική. Αλλά πρέπει να έχουμε τα μέσα να αντιμετωπίσουμε ε, όλους αυτούς τους τομείς και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα σε όλες τις τροπολογίες που αφορούν ε, την ε, γεωργία και οι οποίες, όπως είπατε, δεν μπορούν να ενσωματωθούν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένη και ισχυρή διατύπωση. Και για το 2020 δεν θα ήταν κακό να αναφέρουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δεν έχουμε αναφερθεί σχεδόν καθόλου στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μήπως λοιπόν να ενισχύσουμε λίγο τη διατύπωση εκεί. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η ομάδα μου δεν έχει εκφράσει άποψη, επιτρέψτε μου λοιπόν να το κάνω. Το θέμα της ανεργίας των νέων που είναι μια τραγωδία και η ανάγκη να ξαναδούμε όλα τα μέσα που έχουμε αποφασίσει για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές όπως παραδείγματο χάρη η Γερμανία, η Ολλανδία και η Αυστρία που χρησιμοποιούν συστήματα όπως ε, την μαθητεία των νέων εκεί η ανεργία των νέων είναι ανύπαρκτη σχεδόν. Κάτι τέτοιο λοιπόν ίσως θα έπρεπε να υιοθετήσουμε κι εμείς. Και όταν επισκεφτήκαμε το Λίβανο και την Ιορδανία, μας έλεγαν όλοι ότι οι νέοι θέλουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια ε, και το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης και της λίγο πιο σταδιακής θέλετε προσχώρησης στην τη εκπαίδευση είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε. Έχουμε λοιπόν μέσα, περιορισμένα βέβαια, και οι μαθητευόμενοι όπως ακριβώς και οι φοιτητές θα πρέπει να εποφελούνται από συστήματα και προγράμματα κινητικότητας, ανταλλαγών για περίοδο 6 ή 12 μηνών. Κυρία Μπρεσό, έχετε δίκιο. Η κυρία Μογκερίνη δημόσια μίλησε για την πρωτοβουλία αυτή που αφορά τη μετανάστευση. Βεβαίως και αν θέλουμε να ε, ρυθμίσουμε όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες αυτών των φαινομένων που είναι η πηγή του προβλήματος. Δηλαδή η απόγνωση αυτών των ε, ανθρώπων οι οποίοι εγκαταλείπουν τις χώρες τους και έρχονται στην Ευρώπη. Και αυτό αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι αυτές οι μεταναστευτικές ροές θα τετραπλασιαστούν μέχρι το τέλος του αιώνα. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφήνουμε ανοιχτές πόρτες, περάσματα για τους μετανάστες όπως τη Λιβύη παραδείγματος χάρη. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει σήμερα να περιμένουμε λίγο και θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Μέχρι να μας υποβληθεί το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017. Κυρία Καλπίνιο, θέλετε το λόγο. έτσι ώστε αυτή η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση να μπορέσει να ενσωματώσει και τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση και το θέαμα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι ένα θέαμα αδυναμίας. σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε εντελώς το περιθώριο της ιστορίας. Η κυρία Καλβίνη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώσατε με πολύ βαριές εκφράσεις και ναι, ήθελα λιγάκι να σας πιέσω. Σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μας, τις ευχαριστίες μας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τους εισηγητές. Πραγματικά η προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, μια συμφωνία στο Κοινοβούλιο είναι εξαιρετική. Βρισκόμαστε λοιπόν στη φάση της ε, αναθεώρησης ίσως θα πρέπει να μιλήσω αγγλικά. Μιας και βρισκόμαστε στα μέσα της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης και βέβαια ε, δεν θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε περίπλοκα θέματα από αυτά που συζητήθηκαν σήμερα δεν θα ήταν ορθό να προκαταλάβω τις συζητήσεις για τα ουσιαστικά θέματα που εξήγησαν σήμερα οι αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σημειώσαμε τις ανησυχίες σας και τις αρχικές σας τοποθετήσεις. Χωρίς λοιπόν να προκαταλάβω την συζήτηση επί της ουσίας, να μου επιτρέψετε να κάνω τρεις παρατηρήσεις ως αντίδραση στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που παρακολούθησα. Πρώτα για το γενικό πλαίσιο της τεχνικής μας εργασίας για την προπαρασκευή αυτής της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης. Θα πρέπει να είμαστε διανοητικά ειλικρινείς και έντιμοι. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει αυτή η επανεξέταση. Δηλαδή να επανεξετάσουμε ποια πράγματα αποδίδουν και ποια όχι. Και ε, να φτιάξουμε μια επικαιροποιημένη εικόνα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για περίπλοκη υπόθεση, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της εφαρμογής σε ορισμένους τομείς και ιδίω για τα διαρθωτικά ταμεία. Στην βάση αυτή της αναθεώρησης πια θα κληθούμε να λάβουμε απόφαση εάν θα προχωρήσουμε σε πλήρη αναθεώρηση του ΠΔΠ ή, ή όχι. Γνωρίζω ότι αυτή την διανοητική πειθαρχία την αναγνωρίζει κανείς και στο αρχικό έργο των δύο ε, ε, εισηγητών. Όπως είπε ο κ. Μπέγκε και άλλοι, θα σημειώσουμε θέματα και θα προσεγγίσουμε το θέμα με ιδιαίτερη λογική. Όχι, εξετάζοντας, όχι μόνο εξετάζοντας τα ποσοτικά στοιχεία, αλλά και τα ποιοτικά. Δηλαδή πώς εφαρμόζεται το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι κανόνες εφαρμογής του είναι κατάλληλοι. Θα εξετάσουμε και ενδεχόμενα θέματα που αποτελούν τη γέφυρα για το επόμενο πιδελταπή. Όπως είπατε ορισμένοι εξημών, υπάρχει επίγον χαρακτήρας για την αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων, αλλά ίσως λιγότερο επίγοντα ή λιγότερο όρημα για να ενταχθούν στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Και ίσως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και ποια είναι τα θέματα που θα αποτελέσουν τη γέφυρα για το επόμενο πει. Δεύτερη παρατήρηση, σχετικά με σχόλια που έκαναν οι κύριοι Μαραγάλ, ε, η και και άλλοι, που αναφέρονται στον χώρο των ίδιων πόρων. Η ομάδα των Ευρωβουλευτών που ασχολείται με του ιδίου πόρου γνωρίζετε ότι συνέρχεται τακτικά και εξετάζει διάφορε ιδέε με στόχο να συνταχθεί έκθεση περί τα τέλη του 2016. Θα αποτελέσει αυτό σημαντικό ορόσημο, ξεκινώντα από το Σεπτέμβριο με την διακοινοβουλευτική συνέλευση που θα γίνει στι 7 και 8 Ενάτου, όπου υποθέτω ότι η Επιτροπή σα θα παίξει σημαντικό ρόλο. Χαίρομαι για το γεγονό λοιπόν ότι και το Κοινοβούλιο παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τι εξελίξει αυτέ και εμεί παρακολουθούμε προσεκτικά τι εργασίε τη ε, ε, ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου. Θα εξετάσουμε και άλλα θέματα που μπορούν ε, να θεωρηθούν, όπω είπα, οι γέφυρε για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και εντάσσονται λιγότερο στην τώρα ενδιάμεση αναθεώρηση. Εν τέλει, να έρθω σε ορισμένε από τι ερωτήσει σα σχετικά με ένα ειδικό σχεδιασμό για την Αφρική ή για άλλα σχετικά ζητήματα. Είδα και στον τύπο κάποιες προτάσεις, πράγματα που έχουν προωθήσει κάποιες εθνικές κυβερνήσεις για ένα σύμφωνο για τη μετανάστευση. Η αρχική τοποθέτηση του Πρόεδρου Γιούνκερ ήταν θετική. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Είναι όμως πρόημο να αναμένουμε πολύ συγκεκριμένε προτάσεις σαν αυτές που αναφέρατε. Τούτου εκθετω έχω να κάνω δύο σχόλια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσει εάν μπορεί να αναλάβει περισσότερε δραστηριότητε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων για να αντιμετωπιστούν οι ρίζε του μεταναστευτικού. Επομένω η ΕΤΕ εξετάζει ενδεχόμενες εναλλακτικέ επιλογές, μόχλευση, ξεκινώντας δηλαδή από τα δικά τους κεφάλαια πρώτιστα για να αντιμετωπιστούν οι ρίζες του μεταναστευτικού. Δεν υπάρχουν όμως ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις. Δεύτερο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματιζόμαστε διαρκώς σχετικά με το ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να αντιμετωπιστούν οι ρίζες του προβλήματος της μετανάστευσης. Μιλήσαμε για το Trust Fund για την Αφρική. Επανεξετάζουμε το πώς θα χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα μέσα που μας προσφέρει ο προϋπολογισμός, ο ίδιος ο προϋπολογισμός. Πάλι όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση τουλάχιστον σε σχέση με τα συγκεκριμένα νούμερα που ακούσαμε σήμερα εδώ. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν με συγκεκριμένο τρόπο στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Βεβαίως πολύ ευχαρίστως να επανέλθουμε και να σας εξηγήσουμε τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια πρόταση που θα έχει λάβει σάρκα και οστά εφόσον υπάρξει τέτοια τις επόμενες εβδομάδες. Τελευταία μου παρατήρηση ως εξής σε θετικό πνεύμα. Συνεργαζόμαστε πολύ θετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένω και προσδοκώ συνέχιση τη συνεργασία αυτή τι επόμενε εβδομάδε και μήνε, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το δυνατόν συντομότερο. Ελπίζω δε μέχρι τέλου του έτου. Όπω άλλωστε είπαν και ορισμένοι και των Ευρωβουλευτών σα σήμερα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθύντρια το συμπέρασμά μου από αυτά που είπατε είναι ότι υπάρχει μια θετική συνεργασία. Πολύ ευχαριστώ. Αυτό διότι θα χρειαστεί τέτοια καλή συνεργασία. Με το Συμβούλιο επίσης άλλωστε. Καλώς λοιπόν, ας προσφέρουμε την ενθάρρυνση, όση ενθάρρυνση μπορούμε στους ε, εισηγητές για να προχωρήσουν στην διεκπαιρέωση των συμβιβαστικών με τους ε, σκιώδεις. Εσείς και Όλμπριχτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, λίγα σχόλια. Πρώτα, ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια σχετικά με το έργο μας που όμως ε, ο θετικός της χαρακτήρας οφείλεται στη συνεργασία. Το θετικό του χαρακτήρας οφείλεται στη δική σας συνεργασία. Πρώτα, στην έκθεσή μας δεν αποσκοπούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Ούτε θέλουμε να αντικαταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να κάνουμε εμεί τη δουλειά της. Αυτό που εκφράζουμε είναι η πολιτική θέση του Κοινοβουλίου, τη πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Λέμε δηλαδή τι αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο. Άρα, καταθέτουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και κάποιες προτάσεις για τους τομείς όπου θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θεωρούμε εμείς απόλυτα κατεπίγουσες. Αυτή είναι η βασική τοποθέτησή μας. Δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι που παίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον προπολογισμό και τις τροποποιήσεις του. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση. Δεύτερη, νομίζουμε ότι η ενδιάμεση ή η προσωρινή αναθεώρηση είναι το σωστό χρονικό σημείο για να γίνει επανεξέταση διαφόρων τομέων πολιτικής. Πριν κάνουν την αναθεώρηση αυτή η, της Επιτροπής, οι δικές μας Επιτροπές θα επανεξετάσουν και αυτές όλους αυτούς τους τομείς πολιτικής, της πώληση δηλαδή. Όπως είπε και η Γενική Διευθύντρια, το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι δογματική η τοποθέτησή μας ότι θέλουμε και καλά αναθεώρηση από την αρχή. Έχουμε διεξαγάγει ακροάσεις το αποτέλεσμα ή το συμπέρασμα είναι ότι η αναθεώρηση είναι απολύτως αναγκαία. Αυτή είναι η λογική συνέπεια δηλαδή του έργου που επιτελούμε εδώ. Και νομίζω ότι για να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες, για κάποια θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως η πρωτοβουλία για τους νέους, το ερώτημα είναι υπάρχει αξιολόγηση ή όχι. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό που ο κ. Μάνκα σχετικά δηλαδή με ε, έργα που έχουν υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο. Γνωρίζουμε ότι κάποια από τα έργα αυτά έχουν απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λέγοντας ότι είναι υπερβολικά μεγάλος ο κίνδυνος. Ορισμένοι μου είπαν ότι δεν ε, τους δίνουν χρήματα διότι ούτε το ίδιο το εύση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν του δίνει χρήματα γιατί είναι υπερβολικά ε, υπερβολικό το ρίσκο, το επιχειρηματικό ρίσκο των έργων αυτών. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, για παράδειγμα, του προβλήματος που ανέφεραν οι σοσιαλιστές συνάδελφοί μας. Η διασύνδεση δηλαδή μεταξύ του προπολογισμού του 2017 και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος είναι διαφορετική. Είναι όμω αναγκαίο να καταθέσουμε, να βάλουμε δηλαδή, τα χαρτιά μα όλα πάνω στο τραπέζι πριν από τι διαπραγματεύσει. Δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και να υποχρεώσουμε τον εισηγητή του προπολογισμού του 2017 να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Έχουμε το μήνυμα ότι υπάρχει μια διασύνδεση. Όχι μόνο με αυτό άλλωστε. Υπάρχει και η διασύνδεση με την τακτική προσαρμογή που θα γίνει τώρα με το performance-based budgeting και που πρέπει να δοθεί μια τελική μορφή. Ένα από τα πολύ ευαίσθητα στοιχεία που συζητούμε από την αρχή είναι το πρόβλημα της πολιτικής συνοχής σε σύνδεση με τη μετανάστευση. Ουδής είναι αφελής. Ορισμένες από τις χώρες μέλη επικρίνονται διότι δεν δραστηριοποιούνται και δεν φαίνονται αλληλέγγυες. Ουδής παραπονείται ότι τα χρήματα δεν δαπανώνται. Τα δε, τα δε εθνικά envelopes μπορούν να τα υπερβούν οι χάρες, δεν μπορούν να τα μειώσουν. Μπορούν να προσθέσουν στα εθνικά envelopes, δεν μπορούν να αφαιρέσουν. Είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι το Ταμείο Συνοχής πρέπει να επαναπρογραμματιστεί για να αντιμετωπίσει τον στόχο αυτό της μετανάστευσης. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη μεριά ανοίγουμε ταυτόχρονα την πλησίδα της Πανδώρας. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε δηλαδή ότι τα τα ταμεία και ιδίω συνοχής και τα διαφθορτικά οδηγούν σε μεταφορές πιστώσεων το κοινό στις χώρες μας είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σε αυτά, διότι ανοίγουμε τις αγορές και μια αγορά χωρίς πολιτική συνοχής δεν μπορεί να ανοίξει, παραμένει κλειστή. Ανοίγουμε λοιπόν την αγορά, χρειαζόμαστε όμως την πολιτική συνοχή, συνοχής μάλλον, ως αντιστάθμισμα. Όμως το ερώτημα που τίθεται είναι πού μπαίνει το όριο. Ποιες είναι οι αναγκαίες μεταφορές, που είναι δίκαιες δηλαδή, και πού υπερβαίνει κανεί το όριο. Αυτό όμω είναι συζήτηση για το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Εγώ είμαι Πολωνό. Δεν θέλουμε να αμελήσουμε την πολιτική συνοχή. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να παραλαμβάνουμε διαρκώς να έχουμε κάποιου να μα λένε σας δίνουμε χρήματα και κάνετε αυτά που κάνετε. Ναι, λέμε κι εμεί τότε ότι εμεί προσφέρουμε την αγορά μα. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία. Πάντω αυτή η συζήτηση πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Ίσως αυτό να είναι αντικείμενο συζήτηση για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική. Εμεί είμαστε ευρωβουλευτέ, εκλεγόμαστε. Οι άνθρωποι έχουν, που μα εκλέγουν έχουν ρωτήσει, πρέπει να του δώσουμε απαντήσει. Πάντω δεν είναι αυτή τη στιγμή που θα γίνει αυτή η συζήτηση και επειδή νομίζω όλε και όλοι μα ευχαριστήσατε, θέλω και εγώ να επιστρέψω τι ευχαριστίε για την ε, συνεργασία σα. Ευχαριστώ κύριε Ολμπρίκτ. Ωραία. Σωστή επιλογή Επιτροπή Προϋπολογισμού, γιατί εδώ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα γεγονότα και την πραγματικότητα. Η Ιζαμπέλ, ευχαριστώ. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που διάλεξα την Επιτροπή Προϋπολογισμού, γιατί εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ρεαλιστές. Είμαστε ίσως οι πιο ρεαλιστές μεταξύ όλων των ε, θεσμών και θεσμικών οργάνων και ζητώ συγγνώμη από την Επιτροπή. Εμείς όμως πραγματικά προσπαθούμε να μην εθελοτυφλούμε και να κοιτάξουμε την πραγματικότητα ως έχει. Αυτή η πραγματικότητα είναι προβληματική. Συνεχίζει να είναι προβληματική. Άκουσα την κυρία Μπρεσό και άλλους που αναφέρονται σε αυτό το Ταμείο Συνοχής ε, Συνεργασίας για την Αφρική. Εγώ πολύ θα ήθελα να ενημερωνόμαστε εμείς στο Κοινοβούλιο πριν να ενημερωθεί ο τύπος. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, να οικοδομήσουμε από κοινού κάποιες πρωτοβουλίες γιατί ε, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να είμαστε εμείς ε, ένα σώμα καταγραφής αποφάσεων. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους που με ευχαρίστησαν. Με τις ευχαριστίες σας ε, μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ και τον Γιάνν Όλμπριχτ γιατί με πολύ θετικό πνεύμα εργαστήκαμε μέχρι τώρα. Εμείς θεωρούμε, όπως είπε ο κύριος Σάρουαμά πριν από λίγο, ότι έχουμε πολύ σοβαρές ευθύνες και ότι είναι επίγον να υπάρξουν αποτελέσματα. Αποτελέσματα, σοβαρά αποτελέσματα, βάσιμα και ρεαλιστικά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλα τα μέλη της Επιτροπής που μας στηρίζουν. Νομίζω ότι είδατε ότι έχετε τη στήριξη όλων των συναδέλφων, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι... Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν τελείωσα. Ο κύριος Σαρβαμά έκανε μία ερώτηση. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει δεκτή τροπολογία που να έχει αντικείμενο τη γεωργία. Είπα όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η νομική βάση. Δεν μπορούμε δηλαδή να ανοικοδομήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική. Αν υπάρχει ένα θέμα για επίγουσα στήριξη εν ώψη μιας κρίσης στον τομέα της γεωργίας, βεβαίως αλλά δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε εδώ όλη τη βάση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ναι, ναι, υπάρχουν λύσεις που δεν είναι δημοσιολογικές. Κάποιοι θα τις ονόμαζαν ε, έξυπνος προστατευτισμός. Σίγουρα αυτό θα βελτιώσει πολύ το εισόδημα των γεωργών και ε, δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Βλέπετε λοιπόν ότι έχετε την υποστήριξη όλων των μελών της Επιτροπής, της Επιτροπής Προϋπολογισμού, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα κάνατε μέχρι τώρα. Ακούγοντας όμως αυτά που ανακοινώθηκαν στην ΚΑΠ 21, δεκάδες δις, συν 60 δις για την Αφρική, κάπου όλα αυτά τα ποσά δύσκολα θα μπορέσουν να μεταφραστούν σε πραγματικές πληρωμές. Εν πάση περιπτώσει, στις 28 Ιουνίου το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 θα μας υποβληθεί. Η Κλέρ Μούντι, η οποία δέχτηκε το σημείο που αφορά την έκθεσή της να συζητηθεί στο τέλος της ημερήσης διάταξης, δεν προλάβαμε και επανήλθε. Κλέρ, έχει το λόγο. Thank you, Chair, for your very kind words. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια και ελπίζω να αξίζει την ε, αναμονή. Έχετε την έκθεση για τη Ελπίζω να θεωρείτε ότι είναι μια καλή έκθεση και ότι αναφέρεται στον εξαιρετικό ρόλο που η ΜΚΟ διαδραματίζει. Πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ορισμός, ε, οι εργασίες ε, που γίνονται από αυτές και η δυνατότητα διάδοσης καλύτερων στοιχείων, καλύτερων δεδομένων για το έργο τους. Πρέπει λοιπόν οι αποφάσεις μας να είναι απόλυτα ενημερωμένες Αναγνωρίζουμε επίσης ότι χρειάζεται μεγαλύτερη απλούστευση στον κλάδο αυτόν. Επίσης εναρμόνιση προτύπων και διαδικασιών, παραδείγματος χάρη το διαχείριση συστημάτων στην DG Home τώρα για το θέμα της συχημεροδότησης και τα όρια αυτής. Θα πρέπει να αναφέρετε το όριο το 20% που ισχύει τώρα είναι ένα καλό ποσοστό διότι δεν είναι μόνο μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά είναι και οργανώσει του ε, ιδιωτικού κλάδου. Επίσης ε, το ζήτημα διαγράμματος ε, έχει γι' αυτό ιδιαίτερη σημασία. Το πρόγραμμα πολλές φορές ε, εγκρίνεται με καθυστέρηση και άρα δεν μπορούν πάντα να δαπανηθούν οι πόροι που έχουν χορηγηθεί εντός των χρονικών προθεσμιών. Τέλος, για τις μικρές μη κυβερνικές οργανώσεις που θέλουν να παράσχουν ε, δωρές ε, σε είδος. Τώρα, ε, αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση την οποία ακούσαμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Ο κύριος Γευζόφσκι ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ. Ως και ο δισηγητής του ΕΛΚ πρέπει να κοιτάξω εξαντλητικά, εξονυχιστικά αυτό το ζήτημα. Θέλω ήδη να αναφέρω κάποια ερωτήματα. Πρώτον, τελευταίο συνεδρία του προβλεσμού ψηφίσαμε για τη σύσταση, σύνθεση μάλλον της ομάδας των εμπειρογνωμόνων. Διερωτώμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια διασύνδεση με αυτήν την γνωμοδότηση. Δεύτερον, ένα πιο συγκεκριμένο σχόλιο για το σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνώ με την άποψή σας ότι είναι σημαντικό να έχουμε αναλυτικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι μη κυβερνικέ οργανώσει. Το ζήτημα της διαφάνειας, το θέμα των ε, δικαιούχων, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα πρέπει να καταγράφονται, να καταχωρούνται όλοι αυτοί οι δικαιούχοι. Είτε είναι πανεπιστήμια είτε ιδιωτικέ εταιρείε, επιχειρήσει. Η Κομισιόν συλλέγει μόνο τι προφορίες που είναι απαραίτητε. για κάποιες πληρωμές και οι δικαιούχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τι είδους, οργάνωση εκπροσωπούν. Αν είναι ιδιώτες ε, ή εκπροσωπούν οργάνωση. Κάτι ακόμα για την παράγραφο 5. ότι μπορούμε να χρηματοδοτείτε μέχρι τα 20%. Και βράφω 7 αναφέρεται πως η Κομισιόν θα πρέπει να ελέγξει τη δυνατότητα οι Μικρομείς επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ λαμβάνουν πολλές χρηματοδοτήσεις οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμά τους ATC uh, rather than uh, on individual projects provide and NGOs μιλώ για το ερώτημα εάν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν σκοπό συμβατό με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακολουθούν άλλες πολιτικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σχετικά με τα, όσα είπαμε προηγουμένως. Σχετικά δηλαδή με την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου σχετικά με την έκθεση και πολύ ευχαρίστω να συνεργαστώ μαζί σας για τη σύνταξη του τελικού κειμένου που νομίζω ότι το κείμενο αυτό θα είναι θαυμάσιο. Όπως και ε, το κείμενο που συντάσσουν ο κ. Όλμπερτ και η κυρία Τομά Ευχαριστώ. Άλλος που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Συγχαίρω την Κλέρ Μούντι για την έκθεση και να επιμείνω την ανάγκη της διαφάνειας είναι κάτι το οποίο είδαμε και στις αποστολές που είχαμε στην Τουρκία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία. Φαίνεται πως το έργο θα απλουστευτεί εάν οι εταίροι μας είτε είναι ΜΚΟ είτε κυβερνητικοί θα είχαν, θα είχαν μεγαλύτερη διαφάνεια. Και τέλος οι μικρές ε, ΜΚΟ είναι δύσκολο να καταστήσουμε συμβατές ε, τις μικρές ε, ΜΚΟ με τις βαριές διαδικασίες ε, που εφαρμόζει η Ένωση. Προσβλέπουμε σε μια αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού προκειμένου να ελαφρυνθεί αυτή η διαδικασία. Κατά τη γνώμη σα λοιπόν τι, τι είναι μικρή ΜΚΟ, τι μπορεί να τη διακρίνει, να τη διαφοροποιήσει από μια μικρή που δεν είναι μικρή. Η Κλέρ Μουντή έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τα σχόλιά σας. Βάλατε πολύ ψηλά τον πύχη κύριε Τζεχόφσκι. Σε σχέση είπατε δηλαδή ότι θα συναγωνίζετε την έκθεση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως θα κάνω προσπάθεια για να καταλήξουμε σε κοινή λύση που να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που, που θέσατε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οι τροπολογίες λοιπόν εφόσον προκύψουν θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 35 του πριν από τις 6 το απόγευμα για να είναι παραδεκτές. 15 έκτου συζήτηση, έγκριση της γνωμοδοτήσεως από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ίσως όχι στις 36 έκτου, αλλά ίσως στις 27 έκτου, διότι στις 36 έκτου θα έχουμε μεγάλο φόρτο εργασία γιατί θα έρθει και το σχέδιο προϋπολογισμού για το 17. 15 Σεπτεμβρίου προβλέπεται μάλλον Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου προβλέπεται ε, την τελική ψηφοφορία και μετά στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 2017. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε την ημερησία μας διάταξη. Έχετε άλλα θέματα που θα θέλατε να θίξετε, εάν όχι. Διακόπτω τη συνεδρίαση, η οποία θα συνεχιστεί στις 15 και 16 έκτου. Θα μας λείψει η εργασία της Επιτροπής Προπολογισμών έως τότε. Έρετη συνεδρίαση.